Good morning everybody. Please sit uh, in your... Καλημέρα σε όλους. Παρακαλώ καθίστε για να αρχίσει η συνεδρίασή μας. Buenos días a todos. Καλημέρα σε όλους και όλες. Αρχή η συνεδρίαση της Επιτροπής ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φίλων για σήμερα. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, έγκριση αυτής, την έχετε λάβει. Αν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και συμφωνείτε, θεωρείται εγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Επόμενο θέμα, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 14ης Δεκεμβρίου. Έχετε επίσης την αντίστοιχη ενημέρωση. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτήσει, αλλιώς θεωρούνται εγκεκριμένα και τα πρακτικά. Επόμενο θέμα. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Θα ήθελα να σας ενημερώσω, όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι, ότι στις 3 Μαρτίου θα γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Με εστίαση ιδιαίτερη στο θέμα των ε, προσφύγων γυναικών και μας έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία του στην ε, διοργάνωση αυτή ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου κύριος Μάρτιν Σούλτς και η κυρία Μέρι Ρόμπινσον. Ελπίζω να έχετε όλες την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε αυτή την εκδήλωση την τόσο σημαντική. Ανακοινώσεις Προέδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Έλαβαμε αποφάσεις διαδικαστικές για ορισμένες εκθέσεις, ε, αποστολές και ακροάσεις και θα σας ενημερώσουν οι συντονιστές των πολιτικών σας ομάδων σχετικά. Τέλεια. Προχωρούμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχετε όλοι τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την έκθεση Word, επίτευξη του στόχου κατά της στόχιας δεδομένων των αυξανόμενων εξόδων των οικοκυριών. Έκθεση πρωτοβουλίας ε, με εισηγήτρια την κυρία Τζούλη Ward. Και πάμε αμέσω στην ψηφοφορία. Συμβαστική παριθμόν 3, ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Έχουμε την τροπολογία παριθμόν 37 τώρα. Ψήφι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 η συμβαστική παριθμών 4 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα περάσουμε τώρα στην τροπολογία παριθμών 43 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμό 5 ψήφι Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία παριθμών 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η, συμβαστική, συγγνώμη 50 υπέ κατά αποχές δεν κατάλαβα ακριβώ τι έγινε ηλεκτρονική επαρήθευση παρακαλώ για την 50 ψηφίζουμε τώρα πέρα ή να περιμένουμε λίγο ακόμα ψηφίσατε όλοι ένας ακόμα πέρας Απερίφθη. 14 υπέρ, 16 κατά. Η συμβαστική υπαριθμόν 6 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 82 ψήφι Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 53 ψήφι Κατά αποχές εγκρίνεται ή 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία εγκρινεται η τροπολογια υπάρχει 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική παριθμόν 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66 υπέρ 67 συγγνώμη κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική υπαριθμών 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 68 ψήφι υπέρ. Συγγνώμη, αλλά ε, χύθηκε ο καφές μου. A pesar las mujeres estamos acostumbradas a hacer dos cosas a la vez. Εμείς οι γυναίκες Είμαστε συνηθισμένες να κάνουμε δύο πράγματα ταυτόχρονα. Από ό,τι φαίνεται εγώ δεν είμαι ικανή να πιω ένα καφέ και να κάνω και τις ψηφοφορίες ταυτόχρονα. Φέρτε χαρτιά, δεν φτάνουν.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 Mira, esto cógelo. Sí, pues en una pasta de Ah, voilà. Directamente. A ver. A ver. Nos están grabando. Ορίστε, έχουμε και τηλεόραση και τραβάει πλάνα. Αυτό μας έλειπε. No, si ya me manchamos. Και λεκιάστηκα και από πάνω. Voilà. C'est bon? Está bien? Perfect. Allez. Ahora solo necesito los papeles. Φέρτε χαρτιά, χαρτομάντιλα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε. Η τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν ξέρω αν τα χέρια ή είμαι τόσο χαμένη. Ε, ψηφίζουμε την 68, αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Ένας. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές όχι 76 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83 υπέρ Αποχές συγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος παρακαλώ. γιατί την 85 αρχίζει τώρα η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 13 υπέρ Για να δούμε τι έχουμε εδώ. Έχουν 87 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η τροπολογία 89 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. Η συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία τώρα παριθμονεπτά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 8 υπέρ κατά όχι. Τι όχι. Δεν έχουμε την 8 εδώ τροπολογία. La enmienda 8 de la... Η τροπολογία παριθμών 8, Γκέρικε. Sí, parece que algún grupo tiene la... Τι έγινε. Κάποιο λάθος. Ψήφι υπέρ τη 8, κατά. Άποχες απορρίπτεται. Η τροπολογία 9 ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές γκρίνεται, Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεν έχω καταλάβει τι έγινε. Μπορούμε να ελέγξουμε τη 13 ηλεκτρονικώς, παρακαλώ, άρχιτε ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 14 υπέ. Κατά. Αποχές. Τώρα δεν τολμάω να αγγίξω καφέ. Ευχαριστώ, αλλά θα τα κάνω πάλι. Πού ήμασταν στη 14 είπε; Κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ή 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολόγια 20 υπέρ κατά αποχές ζητώ συγγνώμη 20 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 2 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία παρθμών 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 είπε, κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία 26 είπε κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και περνάμε στην τελική ψηφοφορία έτσι είναι έτσι είναι της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε αρχίζει τώρα ηλεκτρονικά. Εγκρίνεται 18 υπέρ 11 κατά. Συγχαρητήρια κυρία Γουόρντ. Η κυρία Φων Στόρκ ζήτησε το λόγο. Ναι, θέλω να πω κάτι για τα πρακτικά. Ότι θέλω να καταθέσω έκθεση μειοψηφία και ψήφο μειοψηφία. voto particular, ¿no? Es la opinión minoritaria, la de ser quiere depositar después si puede. Si vota contra puede, entonces va a votar contra. Perfecto, pues eh, lo... Μάλιστα. Θα το γράψουμε στα πρακτικά στην ημερήσια διάταξη, λέει η Πρόεδρος. Ε, ψηφίζουμε λοιπόν την επόμενη έκθεση της κυρίας Χάνιμπολ για την κατάσταση των γυναικών προσφύγων και των γυναικών που ζητούν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρχίζει η ψηφοφορία, η τροπολογία 55 ψηφί υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Άποχες απορρίπτεται. Η συμβαστική 5 ψήφι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική παρθμόν 7 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 69 τοπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ 75 διορθώνει η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές χρειάζεται επαλήθευση αυτό γιατί δεν το κατάλαβα ψηφίζουμε την 75 ηλεκτρονικά Πέρασε. εγκρίνεται. Η τροπολογία τώρα υπαριθμών 76 ψήφι Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εδώ έχουμε μια προφορική τροπολογία τώρα. Και έχετε το κείμενο στη λίστα της ψηφοφορίας. Οπότε θα τη ψηφίσουμε αυτή την προφορική τροπολογία. Ψηφί Κατά. Αποχές. Απορρίψετε. Τροπολογία παριθμών 90. Ψηφιπέ Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 91. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 92. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 93. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95. Υπέρ. Κατά Όχι, όχι, έχει καταπέσει, κάνω λάθος, λέει, Πρόεδρος 94. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 134 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 96 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμόν 11 ψήφι υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 105 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Πάμε συμβαστική 12 ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 112 τοπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 113 επέ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 13 ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 14 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 124 περ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 129 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 130 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Παράγραφος 11 σε τρία τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ είναι το αρχικό κείμενο της παραγράφου κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Το τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, 133, τροπολογία σε δύο τμήματα, τμήμα πρώτο υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 135, ψήφι υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 139 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 141 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 143 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 144 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 16 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 174 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 150 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 155 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 156 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 169 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 172 υπέρ. Ορίστε. Κύριε Τι θέλετε, ηλεκτρονική επαλήθευση για ποια, για την 168. Ωραία. Άρχεται η ψηφοφορία. 168. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε. Απερίφθη. 9 ψήφοι υπέρ 18 κατά και μία αποχή. Can I have a check on 169, please? Μπορούμε να ελέγξουμε και την 169, λέει η κυρία Χάνιμπολ. Άντε, ας πάει και 169. Αρχίζει λοιπόν η ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 169. Πέρας. Απορρίπτεται με μία ψήφο διαφορά. Πού είμαστε τώρα. 170 την είχαμε ψηφίσει. Πάμε λοιπόν στην 172. Ψήφι περ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 175. Ψήφι περ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 185 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 188 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 189 υπέρ. Ορίστε. Συγγνώμη. Θέλετε να ελέγξουμε την 188. Ωραία. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 188 αρχίζει τώρα. Πέρασε. Απερίφθη. 11 υπέρ, 17 κατά. Από σφιγμό δεν πάω καλά, από μάτια πάνω κάτω βλέπω. Όχι ότι δεν κάνω λάθη, αλλά κόβει το μάτι μου. Πού ήμασταν? 189 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα δεν κατάλαβα. 190 χρειάζεται ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ. Εγκρίνεται. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι με την ίδια πλειοψηφία, αλλά δεν είναι πολύ σαφές. Τώρα χρειάζεται παλήθευση και για την 191. Ε, λογικό δεν είναι. Ισοψηφία. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 194 σε δύο τμήματα. Τμήμα πρώτο υπέρ. Εν κόντρα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 196 και 197 είναι ταυτόσιμες. Τις ψηφίζουμε μαζί υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 198 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 200 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 203 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 3 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολόγια 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, η 6 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 8 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές αυτό δεν το κατάλαβα πολύ καλά άρα θέλει έλεγχο ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία Περθών 9 αρχίζει η ψηφοφορία Απορρίπτεται. τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική ένα. Έχει και προφορική τροπολογία της εισηγήτριας. Δεν ξέρω αν θέλει να την εξηγήσει. Ναι, να προσθεθεί μια ε, φράση μετά το ε, χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από τη Μεσόγειο ε, για να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 38% ήταν γυναίκες και παιδιά. Εκεί να προσθεθεί. Ενώ η πατερμοστία του ΙΕ για τους πρόσφυγες έχει καταγράψει ότι από τον Ιανουάριο του 2016 τα παιδιά και γυναίκες είναι το 55% όσων φτάνουν στην Ελλάδα για να ζητήσουν άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς είναι για να ενημερωθούν τα στατιστικά δεδομένα. Ελπίζω να συμφωνείτε. Ε... Ναι, ζητώ συγγνώμη. Συμφωνείτε με την ενημέρωση των στοιχείων που μας έδωσε η κυρία Χάνιμπολ για την προσαρμογή αυτή και ψηφίζουμε τη συμβαστική ένα ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές απορρίφεται τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η τροπολογία υπαριθμών 24 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ, κατά άποχες. Δεν κατάλαβα τι έγινε ακριβώς εδώ. Ας το ελέγξουμε. 32 αρχίζει ψηφοφορία. Εγκρίθηκε. Τροπολογία 31 ψήφι υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία παρθών 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 39 σε δύο τμήματα τμήμα πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η τροπολογία τώρα υπαριθμών 40 τι κάναμε την 161 την ψηφίζουμε τη 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 δεν ψηφίζεται διότι κατά πίπτη άρα το ίδιο ισχύει και για την 53 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και τώρα θα περάσουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα Πέρας. Εγκρίνεται η έκθεση 18 υπέρ 10 κατά. Συγχαρητήρια κυρία Χάνιμπολ. ναι, κυρία Στόρχ, θα ήθελα και εδώ να καταθέσω στα πρακτικά ότι καταθέτω ψήφο μειοψηφίας και έκθεση μειοψηφίας. bien, Πολύ ωραία. Τις επόμενες ώρες θα πρέπει να καταθέσετε το κείμενό σας στη γραμματεία, έτσι για να είναι έγκυρη η διαδικασία. Y pasamos a la votación. Και περνάμε στη ψήφιση της απαλλαγής για τον προϋπολογισμό 2014 sobre el presupuesto general de la... Γενικός Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τροπολογία παρθήμου 5, ψήφι Πέ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ. En Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Επαληθεύουμε την 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να σηκώνετε και κανένα χέρι. Ε, δεν ξέρω. Χρειάζεται έλεγχος. Είπαμε από μάτια καλά πάω, αλλά δεν σηκώνετε χέρια. Άρχεται η ψηφοφορία.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 Ισοψηφία. Απορρίπτεται. Και το δεύτερο τμήμα τώρα τι γίνεται. Καταπίπτει πρέπει να το ψηφίσουμε. Πρέπει. Ψήφι υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται και το, το δεύτερο τμήμα, όχι το πρώτο. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 4 υπέρ. Κατά άποχες έλεγχος για την 4 γιατί δεν κατάλαβα τι έγινε Άρχισε ψηφοφορία πέρας απερίφθη τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά αρχίζει τώρα Εγκρίνεται. 22 ψήφοι υπέρ, 6 κατά. Να διαβεβάσετε τα συγχαρητήριά μου στην κυρία Ματέρα. Και πάμε τώρα στην άλλη ψηφοφορία, απαλλαγή 2014 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων. Τροπολογία παριθμών 1, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία παριθμών 2, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 5 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται, 6 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται και πάμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Αρχίζει τώρα. Εγκρίθηκε 22 ψήφοι υπέρ, 5 κατά. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Τελειώσαμε τις ψηφοφορίες.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 Um, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να αρχίσουμε. Έχουμε τρία τέταρτα στη διάθεσή μας. Eh, λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε τρία τέταρτα στη διάθεσή μας για τη συζήτηση αυτή με την κυρία Υπουργό, οπότε καλό θα ήταν να αρχίζουμε σιγά σιγά. Ε, και να ακούσουμε την παρουσίαση της κυρίας Μπούσεμάκε, που είναι Υπουργό Παιδείας Πολιτισμού και Επιστημών των Κάτω Χωρών και ήρθε να μας παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ολλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ήθιστε στην αρχή κάθε εξαμήνου και στην αρχή κάθε προεδρίας να έρχεται ε, να κάνει παρουσίαση του προγράμματος ε, η κάστοτε κυβέρνηση. Ε, την περασμένη εβδομάδα στην Ολομέλη έγινε μια γενική συζήτηση για τις προγραμματικές δηλώσεις τρόπον τεινά της Ολλανδικής Προεδρίας. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω και άκουσα και δικές σας τοποθετήσεις και ερωτήσεις σχετικές με την Επιτροπή μας στη γενική συζήτηση που έγινε για την Προεδρία στην Ολομέλεια. Σήμερα έχουμε την ευκαιρία να εμβαθύνουμε, έχουμε ενώπιον μας την Υπουργό και θα ακούσουμε τα παιδιά και τις ενότητες που σκέφτονται να εμβαθύνουν και να ασχοληθούν ε, από την Ολλανδική ε, Προεδρία. Γεια σας κυρία Μάκερ. καλώς ορίσατε στην Επιτροπή Γυναικών. Θα σας δώσουμε το λόγο και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Παρακαλώ. Αγαπητή κυρία Γκάρσια Περές, θα ήθελα αρχίζοντας να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σήμερα δεν υπάρχουν τόσες πολλές επιτροπές ε, στην Ευρώπη ή συμβούλια όπου εκπροσωπούνται σε τόσο μεγάλο βαθμό οι γυναίκες όπως τη δική σας επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερος που είμαι εδώ. Τον Οκτώβρη πέρσι συναντήκαμε με την κυρία Κασία Περές και συζητήσαμε τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ευρώπη και το πώς επηρεάζουν τις γυναίκες συζητήσαμε για τη σημασία που έχει η δέσμευση στρατηγικού χαρακτήρα υπέρ των ίσων δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Δεν είναι κάτι το αυτονόητο, χρειάζεται διαρκώς να προσδίδουμε τη δέουσα σημασία σε αυτό το θέμα. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της Ολλανδίας θα προσπαθήσουμε να ρίξουμε το βάρος στην ισότητα των δύο φύλων στην Ευρώπη και να προωθήσουμε το σχετικό θεματολόγιο. Προσβλέπουμε στη μελλοντική συνεργασία μαζί σας. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών, Θεωρητικά, σε πολλές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε επιτύχει ισότητα των δικαιωμάτων των δύο φύλων. Όμως χρειάζεται παρακολούθηση, χρειάζεται ενίσχυση αυτών των επιτευμάτων καθημερινά. Χρειαζόμαστε παρεμβάσεις ε, στις τρέχουσες πολιτικές, ακόμη και σήμερα. Τα τελευταία 100 χρόνια, πόρτες που ήταν κλειστές για τις γυναίκες, ε, για αιώνες ολόκληρους, άρχισαν να ανοίγουν μία-μία στην αγορά εργασίας, στο νομικό σύστημα, στα πανεπιστήμια στην πολιτική, ε, στην καθημερινή ζωή, στην οικογενειακή ζωή. Σημαντική κινητήριος δύναμη για αυτά τα επιτεύγματα ήταν η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Στις κάτω χώρε, η μη διακριτική μεταχείριση και η ισότιμη μεταχείριση κατοχυρώνονται στο άρθρο 1 του συντάγματός μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι σαφέστατη ένδειξη για το πώς επωφελούνται καθημερινά οι γυναίκες από τη δουλειά που κάνετε στο Κοινοβούλιο και ειδικότερα εδώ στην Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Παρ' όλα αυτά και πιστεύω θα συμφωνήσετε μαζί μου, δεν αρκεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η νομοθεσία από μόνη της δεν μπορεί να αποτρέψει τα πρόσφατα περιστατικά όπου πολυάριθμες γυναίκες δέχθηκαν σεξουαλικές επιθέσεις, επιθέσεις συγγνώμη, στους δρόμους ε, ευρωπαϊκών πόλεων και πρωτευουσών. Αυτά τα περιστατικά κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και μας υπενθυμίζουν ότι στην πράξη δεν έχουμε επιτύχει ακόμη ισότητα των δικαιωμάτων των δύο φύλων και υπάρχουν νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαρκή προσπάθεια. Αυτό το χρειαζόμαστε περισσότερο από ότι στο παρελθόν. Οι γυναίκες και οι ΛΟΑΔ αγωνίζονται για ίσα δικαιώματα και ισότιμη μεταχείριση εδώ και δεκαετίες με την παγκοσμιοποίηση και με την ε, εισρωή ε, μεταναστών τη σήμερα ημέρα είναι επιτακτική η ανάγκη να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και να μεταφράσουμε σε πράξεις τις ιδέες μας. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις ε, ιδέες και τις αξίες μας ε, σε αυτό το τομέα. Όλοι δεσμεύονται από τις νομοθετικές διατάξεις ε, και τους κανόνες που χαρακτηρίζουν κάθε δημοκρατική κοινωνία. Δεν πρέπει να κλείσουμε τα σύνορα. Θα πρέπει όμως να ε, χαράξουμε σαφέστατα σύνορα. Είναι απαράδεκτη η αδίποτε σεξουαλική βία κατά των γυναικών, όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Η σεξουαλική βία κατά των γυναικών, θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες ε, πληθυσμιακές ομάδες. Σε μία μελέτη, φρά το 2014, μας ενημερώνουν ότι 33% των γυναικών στην Ευρώπη είχαν στη ζωή τους κάποιο τέτοιο βίωμα σεξουαλικής ή σωματικής ε, κακοποίησης. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα νούμερα και θα πρέπει να ασχοληθούμε με την εφαρμογή επιτόπου ε, της κείμενης νομοθεσίας. Έχουμε επιλέξει μία μετριοπαθή μένα στοχευμένη ατζέντα για την Προεδρία των κατοχωρών και βασιζόμαστε σε τρεις προτεραιότητες για την Προεδρία μας μια ένωση που επικεντρώνεται στα βασικά που δημιουργεί ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας μέσω της καινοτομία και που με ενεργό τρόπο οδηγεί σε ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στην κατάρτιση της πολιτικής. Η Προεδρία μας θα θέσει στην μερίσια διάταξη ε, των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου πολλά ζητήματα που σχετίζονται με την ισότητα ε, των δύο φύλων. Τους επόμενους έξι μήνες λοιπόν θα συζητηθούν πολλές ε, σχετικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα γίνουν διαπραγματεύσεις για πολλές από αυτές τις πρωτοβουλίες, όπου και συνιστά μεγάλη πρόκληση. Είναι λοιπόν μεγάλο το έργο που μας περιμένει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και θα προσπαθήσουμε με ειλικρίνεια να συμβάλλουμε ε, ώστε να καταλήξουμε συμβαστικές λύσεις ε, για τις εκκρεμείς οδηγίες. Αναλαμβάνουμε δέσμευση να προωθήσουμε τις συζητήσεις ε, για την οδηγία για την ισότιμη μεταχείριση καθώς και την πράξη για την προσβασιμότητα. Επίσης, ε, θα διευκολύνουμε μια παραγωγική συζήτηση στην ε, ομάδα υψηλής εργασίας, ε, υψηλού επίπεδου, συγγνώμη, για το gender mainstreaming, την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των δύο φύλων, δηλαδή στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίσαμε την περασμένη εβδομάδα στο Άμστερνταμ. Ε, εκπροσωπήθηκαν όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ε, με, ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας που καταφέραμε στην ομάδα υψηλού επίπεδου να συγκεντρώσουμε εμπειρογνώμονες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόλις άρχισε το 2016 θα υποστηρίξουμε το ύπατη εκπρόσωπο αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς μια ισχυρή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την 60η Σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για το καθεστώς των γυναικών και προς βλέπουμε φυσικά και στην δική σας συμμετοχή. Επίσης, ισχυρή δέσμευση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 1325 ε, για τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια. Το Μάρτι η Προεδρία της Ολλανδίας ε, θα, προ... θα εισηγηθεί σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ βασιζόμενη ε, στην παρουσίαση των πρωτοβουλίων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των δύο φύλων και το σχέδιο δράσεων για την ισότητα των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤ. Θα ήθελα επίση να υποφεληθώ τη σημερινή ευκαιρία για να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων για την εξαιρετική δουλειά που κάνει χωρί τα κατάλληλα δεδομένα και την έρευνα. Δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά την πολιτική μα. Βλέποντα τελευταία επικαιροποίηση του δίκτυ ισότητα των δικαιωμάτων, μπορούμε μόνο να συμπεράνουμε πω μα περιμένει ακόμη μακρύ δρόμο στην Ευρώπη. Ε, Στι έξι τομεί, ε, ε, εργασία, χρήματα θέματα γνώσης, ε, χρόνος, ε, ισχύς και υγεία, βλέπουμε ότι ε, εξακολουθεί να υπάρχει το χάσμα ανάμεσα στα δύο φύλλα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα σας δώσω συγκεκριμένα νούμερα εν είδη παραδείγματος. Παρότι η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι ελαφρά υψηλότερη στην Ολλανδία σε σχέση με άλλες χώρες, σε μόνο 53 γυναίκες είναι οικονομικά ανεξάρτητες, μόνο 53%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το ίμιση των γυναικών στις κάτω χώρες αδυνατούν να ε, κερδίσουν τα προστοζήν. Αυτή η κατάσταση με ανησυχεί. Ανησυχώ, διότι πιστεύω ότι η οικονομική ανεξαρτησία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για την αυτονομία στην, ε, στην ύπαρξή μας. Η Σιμών Ντομποβουάρ εντόπισε αυτόν τον τομέα ως ε, μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις ε, των γυναικών για να χειραφετηθούν. Και την δήλωση ε, το, του τρίου των τριών χωρών γύρω από την Προεδρία για την ε, ισότητα των γυναικών που συνέταξα μαζί με τους συναδέλφους από τη Μάλτα και τη Σλοβακία και που ε, προσυπέγραψαν τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ στις 17 ε, Δεκεμβρίου. Διαπιστώνουμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η διάσταση διότι μόνο έτσι μπορούμε να αυξήσουμε την αποσχολησιμότητα των γυναικών και να μειώσουμε τον κίνδυνο της στόχιας και του κοινωνικού αποκλείσμου. οικονομική ανεξαρτησία επίσης κάνει αθεκτικότερες ε, τις γυναίκες ε, και επίσης ε, αξιοποιούν χάρη στην οικονομική ανεξαρτησία τις δεξιότητες τους, δεξιότητες που είναι αποφελείς για τις ίδιες αλλά και εν γέννη για την κοινωνία. Οι οικονομικά ανεξάρτητες γυναίκες μπορούν να κάνουν ε, με ανεξάρτητο τρόπο τις επιλογές τους ε, και η εξασφάλιση της οικονομικής ανεξαρτησίας ε, μπορεί έτσι να συμβάλλει στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών. Εάν μια γυναίκα έχει επαρκείς οικονομικούς πόρους για να φροντίσει την ίδια και την οικογένειά της, ε, τότε νομίζω ότι ίσως το βρει, ε, μπορεί ευκολότερα να ε, εγκαταλείψει κάποιον σύντροφο που την κακοποιεί. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής, η οικονομική χειραφέτηση ισοδυναμεί με πραγματική ανεξαρτησία. Δεν είναι μόνο ο οικονομικός παράγοντας ε, και Υπάρχει ο γύρος της χειραφέτησης ε, ε, στις κάτω χώρες. Ποιος είναι ο στόχος αυτή τη της είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση για τη σημασία τη οικονομική ανεξαρτησία. ενθαρρύνοντα έτσι τις γυναίκες να συμμετέχουν ε, στην αγορά εργασία ε, για να γίνουν πιο ανεξάρτητε ε, και για να έχουν μια κρατιότερη θέση στην κοινωνία. Ε, όσο κάναμε αυτόν τον γύρο στην Ολλανδία, μίλησαμε με δεκάδες ε, γυναίκες ε, και καταλήξαμε σε συμφωνίες με πάρα πολλές επιχειρήσεις, δήμους και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Χάρη σε αυτές τις συμφωνίες υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και δημιουργούνται περισσότερε δυνατότητε για τι γυναίκε. Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 1.800 γυναίκε ε, συμμετείχαν σε τέτοιε εκδηλώσει που εντάσσονται στο γύρο τη χειραφέτηση ε, σε όλη την επικράτεια τη χώρα, ε, συζητήσει για την οικονομική ανεξαρτησία, χρήση των δεξιοτήτων, των ταλέντων που έχουν οι γυναίκε, αξιοποίηση ευκαιριών, ανεξάρτητε επιλογέ. Έκαναν πάρα πολύ γενναία βήματα σε οι σχεδόν 2.000 γυναίκες και είμαι περήφανη για αυτό. Με αυτό το γύρο τελικά καταλήξαμε ε, σε πλούσια βιώματα τα οποία χρησιμοποιούνται και ως πρακτικές για γυναίκες ε, που κατέκτησαν την οικονομική ανεξαρτησία και μπόρεσαν ε, να αξιοποιήσουν τα ταλέντα σου. Η Ραχάντ Ελκαμπή, παραδείγματος χάρη, τη συνάντησα προσωπικά. Είναι η Ιρακινής προέλευσης και μεγαλώνει μόνη στα τέσσερα παιδιά της. Όταν ε, πήρε διαζύγιο, έπρεπε να αρχίσει να δουλεύει και πήγε σε μια ε, εταιρεία που λέγεται Van Halley. Εκπροσωπήθηκε και στον Ταβός η εταιρεία αυτή την περασμένη εβδομάδα. Ε, παράγει μποξεράκια ε, για γυναίκες και για άντρες από παλιά τη shirts. Έκανε μια, ένα σεμινάριο στη συνέχεια για μαγειρική και κατέληξε στην Ακαδημία για Επιχειρηματίες όπου ε, άρχισε ένα μάθημα για την επιχειρηματικότητα με 10 ταλαντούχες γυναίκες ε, και ε, για τη Ραχάτε ήταν ένα σημαντικότερο βήμα για να εκπληρώσει τα όνειρά της και άνοιξε το δικό της εστιατόριο και πολύ θέλω να πάω μια μέρα. Είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για το τι σημαίνει εκπαίδευση, κατάρτιση και οικονομική ανεξαρτησία για τις γυναίκες. Σε κάτι διάρκεια αυτού του γύρου χειραφέτης, με αυτές τις ιστορίες όπως αυτή τη Ρακάτε, με κάνουν να συνειδητοποιήσω ότι δεν γίνεται όλα να τα προβλέψουμε στη ζωή. Μπορεί να λήξουν οι σχέσεις, χρειάζονται τα παιδιά φροντίδα, μπορεί ο σύντροφος να χάσει τη δουλειά του και χάρη σε αυτές τις πρωτοβουλίες χειραφέτησης μαθαίνουν να επενδύουν στον εαυτό τους οι γυναίκες να κατακτούν την ανεξαρτησία τους. Ελπίζω να σας εμπνεύσει και σας αυτό το παράδειγμα. Θέλω να μοιραζόμαστε τα βιώματα μας, τις ιστορίες, τις εμπειρίες που έχουμε σε, επίπεδο, ε, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να σημειώνουμε διαρκώς πρόεδρο. Θα ήθελα ε, εν κατακλείδη να τονίσω ότι κατά τη γνώμη μου η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένας αξιόπιστος και αποτελεσματικός τρόπος ε, για να καταλήξουμε συμβαστικές λύσεις ε, με τα 28 κράτη-μέλη και ε, σε διαθεσμικό επίπεδο με το Συμβούλιο και τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Όπως είδαμε και στον λόγο του Προέδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, η κυβέρνηση των κάτω χωρών θα εντατικοποιήσει τις σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας τους, ε, ούτως ώστε με βιώσιμο, συστηματικό, στρατηγικό τρόπο να συνεργαστούμε με ένα δημοκρατικό όργανο που έχει τόσο κέρια σημασία για την νομιμοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ξαναλέω αγαπητά μέλη της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Πιστεύω στην ανταλλαγή γνώσεων, στο να μαθαίνουμε μαθαίνουμε από τις εμπειρίες των άλλων. Μόνο έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε τις πολιτικές μας και να είμαστε αποτελεσματικότεροι στις προσπάθειες που κάνουμε για την υλοποίηση των στόχων μας. Ας ενισχύσουμε τις προσπάθειες που κάνουμε, ούτως ώστε η διάσταση ισότητας των δύο φύλων να κερδίσει έδαφος στην Ευρώπη. Αυτό είναι ο σωστός τρόπος να αρχίσουμε με ανταλλαγή των απόψεων και των βιωμάτων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Muchas gracias, eh, señora Busenmarker. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπούσεμακερ. Θα έχουμε ένα πρώτο γύρο τοποθετήσεων σε επίπεδο συντονιστών πολιτικών ομάδων και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Σας παρακαλώ να τηρείτε αυστηρά το χρόνο αγόρευσή σας για να μπορέσουν να μιλήσουν όλοι. Από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα η κυρία Λεγκρίπ έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς Υπουργέ που ήρθατε σήμερα εδώ για να παρουσιάσετε τις αντρές γραμμές της Προεδρίας σας και τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει για μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ευχαριστούμε που αφιερώνει το χρόνο σε αυτή τη συζήτηση για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα τις κατοχώρες, μπορώ και εγώ να καταθέσω τη μαρτυρία μου αν και το είπατε. Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που εδώ και πολύ καιρό δίνει μεγάλη έμφαση την επίτευξη και την πλήρη εκδίπλωση των ε, ταλέντων και των ιδιαίτερων δεξιοτήτων των γυναικών και στην ε, πραγματική υλοποίηση της ισότητας ανδρών και γυναικών. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαρκής Ολλανδική στράτευση από το σκοπό, ε, η οποία είναι και παλιά, να ανθίσει και κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας και να δώσει καλά αποτελέσματα πείθοντας τους συναδέλφους γύρω από το τραπέζι των στο Συμβούλιο. Και ένα άλλο χαρακτηριστικό που αναγνωρίζουμε συχνά στις κατοχώρες για πολλά θέματα είναι ο πραγματισμός σας και η αποτελεσματικότητά σας. Ελπίζουμε λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά να αξιοποιηθούν και όντω να αξιοποιηθούν για το σκοπό της μεγαλύτερης ισότητα ανδρών και γυναικών. Από την πλευρά του ΕΛΚΑ έχουμε βεβαίως κάποιε προτεραιότητες και αρκετέ ε, μέρημνες και σας ευχαριστώ που τα σχολιάσατε εκτενώς και από την αρχή της ομιλίας σας όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, ασχέτως τόπου, συνθήκων, ομάδων πληθυσμού που μπορεί να είναι υπεύθυνε, διότι έχει διαπιστωθεί αύξηση της μορφής βίας κατά των γυναικών. Και μάλιστα μαζικής παρενόχλησης, πρόσφατες μορφές που ανησυχούν ιδιαιτέρως τους πολίτες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η Προεδρία σας θα ασχοληθεί σοβαρά με την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και ότι θα εντείνουμε τις ε, προσπάθειές μας και τον αγώνα μας. Ως ΕΛΚ είμαστε πραγματικά αφοσιωμένοι Την προσπάθεια που θα πρέπει να κάνουμε ως Ευρωπαϊκό Θεσμικό Όργανο για την υλοποίηση των ισχυών των ευρωπαϊκών κανόνων. Χρειάζεται περισσότερη ε, δραστηριοποίηση να υποδαβλίσουμε λίγο την ε, καθημερινή δράση του καθενός για να υπάρχει ορθή εφαρμογή ώστε το πλαίσιο και οι κανόνες που ήδη παρέχουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να φέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Επίσης, ε, μας ενδιαφέρει ο σεβασμός της αρχής της επικουρικότητας, γι' αυτό και αυτές είναι οι αδρές γραμμές, οι βασικές ε, προτεραιότητες, τις οποίες θα παρακολουθούμε στην ε, διάρκεια της Προεδρίας σας, την δική σας δράση. Θα υπάρχει αρκετή πίεση Ευχαριστώ πολύ. Θα σας παρακαλούσα να ορίσουμε χρόνο αγόρευσης. Ένα δίλεπτο για να μπορέσουν όλα να μιλήσουν. Η κυρία Ρενά, εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ για την ομιλία σας. Ευχαριστώ και για τα σχόλια για την μαζική βία. Προσωπικώς έχω σοκαριστεί ιδιαίτερος όταν συσχετίζεται αυτού του είδους η βία με την μετανάστευση. Βρίσκω ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνοι αυτοί οι συσχετισμοί όταν τα βλέπουμε από αυτή την προοπτική. Για μα η ισότητα πρέπει να είναι προτεραιότητα όχι μόνο όταν υπάρχουν ιδιαίτερα γεγονότα που φαίνεται να την απειλούν, διότι έχουμε πολλά τέτοια επεισόδια εδώ και πολλά χρόνια. Και στη διάρκεια του χρόνου μόνο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα στερεότυπα. Αυτά ακριβώ τα στερεότυπα προκαλούν μορφέ βία κατά των γυναικών. Το πρώτο ερώτημα που έχω να θέσω είναι πώς σκέφτεστε ως Προεδρεύουσα να υπερασπιστείτε το δικαίωμα διάθεσης του σώματος των γυναικών, διότι είναι και αυτό το ζήτημα. Πώς μπορούμε να θεσπίσουμε πολιτικές που επιτρέπουν στις γυναίκες να διαθέσουν όπως θέλουν το σώμα τους, και εδώ αλλά και αλλού Λόγω χάρη θέλουμε να ε, προβλέψουμε στα αναπτυξικά μας προγράμματα συγκεκριμένες δράσεις εκπαίδευσης ε, για να μπορέσουν οι γυναίκες να έχουν πρόσβαση και ε, αντίληψη των στοιχείων αυτών, της διάθεσης του σώματος και της αντισύλληψης για παράδειγμα. Ε, όλες οι μορφές της βίας. Ε, τώρα τα στατιστικά, τα στατιστικά δεδομένα. Μια γυναίκα μια στι τρει γυναίκε είναι θύμα είτε ψυχολογική είτε σωματική βία. Με τέτοιου είδου στατιστικά στοιχεία, τι κάνουμε για να υποχρεώσουμε τα κράτη να κυρώσουν τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Σω είναι ένα θέμα που θα μπορούσατε να θέσετε σε επίπεδο συμβουλίου για την υλοποίηση τη σύμβαση αυτή. Και έπειτα το δικαίωμα τη οικονομική ισότητα. Αυτό το δικαίωμα δεν υπάρχει. Υπάρχει διακριτική μεταχείριση στον χώρο τη εργασία, το μισθολογικό, ε, στις, στα επιδόματα. Πώ το Συμβούλιο μπορείτε να καταρτήσετε μια πραγματική στρατηγική για να πάψει αυτή η οικονομική διακριτική μεταχείριση. Επίση, το δικαίωμα συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου. Υπάρχει ένα οδικό χάρτη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να προβλέψετε και μια άδεια πατρότητα και να την προθέσετε στο Συμβούλιο για να υπάρχει καλύτερο συσχετισμό, μάλλον καλύτερη ε, σχέση με την ισορροπία που μπορεί να έχει κανεί με τον ε, σύντροφό του και τι συμφωνίε επαγγελματικού οικογενειακού βίου. Και για τι ε, γυναίκε στα δικαιωτικά συμβούλια, για τον βίο των επιχειρήσεων, για να το πούμε έτσι. Έχουν γίνει πολλέ συζητήσει εδώ και μάλιστα είναι θέματα που συζητώνται εδώ και χρόνια αυτά. Αλλά δεν έχουν δώσει κάποια συγκεκριμένη έκβαση. Δεν πρέπει να υπάρξει πολιτική βούληση από όλε τι πλευρέ για να καταφέρουμε κάτι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Από του Πρασίνου. Η κυρία Ρέτκια. Sorry. Ε, first, ε, first. Ε. Συγγνώμη. Προηγουμένως η κυρία Νιτφέλτ από τους φιλελευθέρους με τη σειρά οι πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Καλώς ορίσατε Υπουργέ Μπουσιμακέρ στα Ολλανδικά η κυρία Νιτφέλτ. Καταρχάς θα ήθελα να σας εκφράσω τον προσωπικό μου σεβασμό και να σας πω πόσο σας τιμώ για τα όσα κάνετε στις κάτω χώρες και ελπίζουμε και για την Ευρώπη το επόμενο εξάμεινο. Τις τελευταίες εβδομάδες κάποια στιγμή σκέφτηκα πω πω τι φανταστικά νέα από την κολονία και μετά γνωρίζουμε ότι όλοι έχουν γίνει φεμινιστές στην Ευρώπη, σέβονται τις γυναίκες, γνωρίζουν ε, ότι όταν λες όχι σημαίνει και όχι. Τι φανταστική εξέλιξη αυτή. Δυστυχώς τα πράγματα έχουν κάπως διαφορετικά στην πραγματικότητα. Δεν είναι όλοι φεμινιστές. Και μάλιστα ουδέν νεότερο από το δυτικό μέτωπο. Το είπατε κι εσείς μια γυναίκα ε, στις τρεις ε, απέχει πόρο από όλα αυτά. Ξέρει τι σημαίνει και βιασμός και σεξουαλική παρενόχληση και βία. Δείχνει μια δημοσκόπηση της Eurostat ε, ότι 52% ε, των πολιτών θεωρούν ότι μια γυναίκα που έχει μείνει φούστα και κυκλοφορεί στο δρόμο προκαλεί. Και ότι αρχίζουν να φοβούνται οι γυναίκες να πάνε μόνες τους να πιούν κάτι. Ε, αυτά που έγιναν στην κολονία είναι αποτρόπαια, είναι φρικτά και αποκρουστικά, αλλά ε, υπάρχει βία κατά των γυναικών και ο σεξισμός που είναι το πρώτο βήμα για τη βία κατά των γυναικών και θα πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά στις προτεραιότητες. Εμένα με εκπλήσει το γεγονός ε, ότι στις 7 Δεκεμβρίου το τρίο της Προεδρίας, οι τρεις επόμενες Προεδρίες δηλαδή, ούτε καν το αναφέρουν αυτό. Μετά από αυτά τα γεγονότα της κολονίας θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει ε, και να καταλάβουμε ότι είναι ένα φαινόμενο που πρέπει να μας απασχολήσει. Υπάρχουν χώρες που θέλουν να κάνουν μαθήματα τώρα, λέει, στους ετούντες άσυλο για το πώς ε, σεβόμαστε τις γυναίκες και τους ομοφιλόφιλους στην Ευρώπη. Μπράβο, ωραία μαθήματα. Να κάνει φροντιστήριο και η καθολική κυβέρνηση, ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η πολωνική κυβέρνηση και πάει λέγοντας. Ωραία είναι αυτά τα ιδιαίτερα που θέλουν να τους κάνουν, αλλά να πω ότι ε, είμαι έξελη από κάποιο ευκαιριακό και συγκυριακό φεμινισμό, από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα για το τι σημαίνει να σέβεσαι τις γυναίκες, αλλά που το χρησιμοποιούν τώρα δημαγωγικά και λαϊκιστικά για να εξυπηρετήσουν τη δική τους ρατσιστική ατζέντα και εγώ που είμαι φεμινίστρια δεν θέλω ούτε να τους ξέρω. Και δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Μιλήσατε για την οριζόντια οδηγία. Θα πρέπει να λήξει αυτή η προσπάθεια μέσα στο εξάμεινο, διότι τραβάει χρόνια. ΛΟΑΔ, ο δικός χάρτης, θα είμαστε ευγνώμονε αν το καταφέρει αυτό η Ολλανδική μα Προεδρία και το πιέσει, διότι με την επόμενη Προεδρία που είναι η Σλοβακική, χαιρετίσματα δεν το θόλου. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη από την Ολλανδική κυβέρνηση. Προσωπικά κάπως απογοητεύτηκα εγώ από το ισχνό αποτελέσματα, τα ισχνά αποτελέσματα του προγράμματος, σε πάση περιπτώσει, και ως μέλος του κόμματος D66 των ε, φιλελευθέρων ε, των αριστερών ε, στην Ολλανδία. Θέλω να σας ρωτήσω τι λέτε για τις μονογονικές οικογένειες ή για τις γυναίκες που ζουν μόνες τους, τον οικοκυριό του ενός προσώπου που συχνά είναι γυναίκες και είναι το 1 τρίτο των οικοκυριών. Έχετε καμιά μέρημνα γι' αυτό. Ευχαριστώ. Τώρα έχει το λόγο κυρία Ρέτκε. Okay. Ευχαριστώ, θα τον λάβω. Ευχαριστώ κυρία Ουσμάκερ που ήρθατε. Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να ε, έχουμε διάλογο. Θα επικεντρωθώ σε ένα μόνο σημείο, διότι πιστεύω ότι μπορείτε σε αυτό το τομέα να κάνετε ακριβώς τη διαφορά και να δώσετε μια όθηση από τη δική μου τη Σκόπια έχει παραγκονιστεί πιστεύω το θέμα αυτό και είναι ακριβώ το θέμα των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια. Ξέρετε ότι από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει αρκετή ε, απογοήτευση, διότι δεν έχει δοθεί αρκετή προτεραιότητα ω τώρα, όσο θα ήθελε τουλάχιστον η, δική μα Επιτροπή και το ίδιο είδαμε και με την οδηγία για την ε, άδεια Δεν ε, έχει προχωρήσει και Μπορεί μάλιστα να περιοριστούν ακόμη περισσότερα αυτά τα δικαιώματα από άλλε οδηγίε. Πιστεύουμε σε αυτή την Επιτροπή ότι δεν θα έπρεπε να έχει την τύχη τη οδηγία τη άδεια πατρότητα και η οδηγία για τι γυναίκε στα διοικητικά συμβούλια. Υπήρξαμε πολύ φιλόδοξοι στην πρόθεση του θέματο αυτού και προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το τέλμα που είχε φτάσει να έχει, στο οποίο είχαν καταλήξει οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε λοιπόν να δοθεί μια νέα όθηση για να πετύχει ο οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη, υπάρχει απαραίτητη πολιτική βούληση και ελπίζουμε ότι στη δική σας Προεδρία θα καταφέρετε να κάνετε κάτι σχετικά και να φέρετε τη διαφορά. Ευχαριστώ πολύ. Από την ΚΟΕ, η κυρία Ευχαριστώ και εγώ πολύ γρήγορα να θίξω κάτι που ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Τα γεγονότα στην κολονία και η συζήτηση που ακολούθησε. Ως φεμινίστρια αισθάνομαι ότι οι ρατσιστικές εκδηλώσεις που είδαμε ε, εκμεταλλεύονται το θέμα αυτό για να προωθήσουν τι δικέ του αξίε, λέγοντα ότι του ενδιαφέρουν τα δικαιώματα των γυναικών και θέλουν να προστατεύσουν τα σώματά μα. Εμένα πραγματικά με προσβάλλει αυτό στο μηνύστριο. Θα πρέπει να είμαστε σαφεί για το ότι υποκρύπτει κάθε τέτοια πρόθεση και ποιοι υπερασπίζονται πραγματικά τι γυναίκε. Μιλάμε κυρίως για μια σοβινιστική νοοτροπία και σοβινιστική κυριαρχία εδώ. Ε, το έχουμε αυτό και στη Σουηδία, στην σουηδική νοοτροπία άλλωστε. Κάτι άλλο ε, που θέλω να καλωσορίσω είναι ότι θα εργαστείτε για το θέμα της οικονομικής ανεξαρτησίας, το βρίσκω άκρος, ιδιαίτερα σημαντικό και το θέμα της ε, ισότητας και της ε, πρόσβασης των ΛΟΑΔ είναι επίσης σημαντικό, θα έχει μεγάλη διαφορά για πολλές γυναίκες εάν πετύχει. Από την άλλη, νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε στα δικαιώματα των γυναικών συγκεκριμένα. από την οπτική γωνία των γυναικών στην Ευρώπη έχουν την αίσθηση ότι έχει φτάσει σε αδιέξοδο η δουλειά για την ε, πρόθεση της ισότητας ε, στον εργασιακό χώρο. Δεν υπήρχαν σημαντικέ κινήσεις τα τελευταία πέντε χρόνια. Οι αδιαπατρότητα και αδιαμετρότητα στις προτάσεις αποσύρθηκαν. Θα θέλαμε κάτι να αντικαταστήσει αυτές τις προτάσεις σε σχέση με τις άδειε που να είναι τουλάχιστον ουδέτερε ω προ το φύλλο από τη δική μα την οπτική γωνία, αυτό θα ήταν το ιδανικό, και να ενισχύσουμε τα εργασιακά δικαιώματα των γυναικών. Όχι μόνο στη θέση των ε, διοικητικών συμβουλίων ή στι ε, ηγετικέ θέσει των επιχειρήσεων. Πρέπει να ενισχυθούν οικονομικά οι γυναίκε και όταν είναι απλέ εργαζόμενε. Και Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα τη δική σας στενή συνεργασία για να ζητήσουμε μια νέα στρατηγική για την ισότητα των γυναικών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Χωρίς την απαραίτητη πολιτική βούληση δεν ξέρω πώς θα προχωρήσουμε την επόμενη πενταετία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τα πράγματα και δεν ξέρω πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε ζητήσει τη στρατηγική αυτή από το σώμα μας, αλλά πρέπει η δουλειά μας να προχωρήσει. Θέλουμε να δείξουμε στις γυναίκες στην Ευρώπη ότι τη δουλειά αυτή, την, ε, τις πεντατές αυτές τις παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη και ότι έχουμε και την πολιτική πρόθεση να τα προωθήσουμε. Γι' αυτό ευχαριστώ και τους συναδε... συναδέλφους που έχουν λάβει πρωτοβουλίες για την ε, καταπολέμηση των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κορίτσιων και ιδίως την κύρωση της Σύμβασης του Κωνσταντινούπολου. Ευχαριστώ. Ε, <clears throat> λοιπόν, για να κλείσουμε με τους συντονιστές θα δώσουμε το λόγο στην Υπουργό για να απαντήσει και αν έχουμε χρόνο στη συνέχεια θα ακολουθήσουν και άλλες τοποθετήσεις από τα υπόλοιπα μέλη. Α, κυρία Γιούτο, είχατε ζητήσει το λόγο. Συγγνώμη, δεν σας είχαμε δει. Παρακαλώ, η κυρία Γιούτο έχει το λόγο. Κανένα πρόβλημα, ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα να ευχαριστήσω τον Υπουργό Μπουσμάκερ που είναι εδώ Να πω απλώς ότι πριν από έξι μήνες όταν ξεκίνησε η Προεδρία του Λουξεμβούργου και πάλι ακούσαμε τότε μια παρουσίαση που ανακοίνωνε μια σειρά από πρωτοβουλίες με αρκετό ενθουσιασμό και αργότερα είδαμε απέναντίας να αποσύρεται η πρόταση για την άδεια μητρότητας Είδαμε για πρώτη φορά το ευρωπαϊκό έτο που θα έπρεπε να είναι ευρωπαϊκό έτο για την καταπολέμηση των ομοσπονδίων κατά των γυναικών και είδαμε και πώ ξεκίνησε η φετινή χρονιά, το 2016 με τα γεγονότα τη Κολονία. Δεν έγινε λοιπόν ακριβώ αυτό και πέραν των καλών προθέσεων στο επίπεδο τη πράξη. Το μεγάλο πρόβλημα τη ανεργία των γυναικών α πούμε. Και σε σχέση με όσα είπαν και οι συνάδελφοι πώς σκοπεύει η Ολλανδική Προεδρία να ε, καλύψει το θέμα αυτό που ξέρουμε ότι είναι διαρθρωτικό. Τις προάλλες ήρθε για μία ακρόαση στην Επιτροπή Απασχόλησης ο Υπουργός Οικονομικών της Ιταλίας για να παρουσιάσει ένα νέο πρόγραμμα, μια ρύθμιση για να καλύψει προσωρινά το πρόβλημα της ανεργίας στην Ευρώπη, ένα γενικό πρόγραμμα. Όμως η ανεργία των γυναικών από την δική του την γωνία δεν περιλαμβανόταν, δεν καλυπτόταν από αυτήν την συλλογική, από το συλλογικό ελιγμό που έγινε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, τα κράτη-μέλη πώς ασχολούνται λοιπόν συγκεκριμένα με το πρόβλημα της ε, γυναικείες ενεργείες. Το επίπεδο του Συμβουλίου μάλιστα, ως Ιλλανδική Προεδρία σκοπεύετε να προβλέψετε κάποια μέτρα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη του Συμβουλίου για να προσπαθήσετε να υλοποιήσετε στην πράξη κάτι που πραγματικά να ωφελήσει τις γυναίκες αυτές που περισσότερο κινδυνεύουν από την ένδια. Ε, δεν μιλώ μόνο για αυτές που έχουν χάσει την δουλειά τους. Το ανέφερε και η συνάδελφος στην παρέμβασή τη. Ευχαριστώ κύριε Γιώτο. Τώρα έχει το λόγο για να κλείσει η συζήτηση υπουργό και ζητώ συγγνώμη από του συναδέλφου που ζήτησαν το λόγο, αλλά δεν θα προλάβουμε. Σίγουρα θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε τις ερωτήσεις σας γραπτός. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι παραπάνω, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα η Προεδρία να σας απαντήσει. Παρακαλώ, Υπουργέ, έχετε το λόγο. Um, Ευχαριστώ. σχολιάσατε όλοι σημαντικότατα ζητήματα και είμαι σίγουρη ότι θα προκύψουν με κάποιο τρόπο όλα αυτά τα θέματα που εγείρατε κατά τη διάρκεια της ε, Προεδρίας. Κυρία Λεγκρίπ, γνωρίζω την ισχυρή σας δέσμευση ε, και γνωρίζετε και εσείς τη δική μας στο παρελθόν και στο μέλλον σας διαβεβαίω θα αγωνιστούμε για να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση ε, σε σχέση με τις γυναίκες. Είστε αποτελεσματικοί και σας χαρακτηρίζει ο ρολισμός, όπως και όλες τις γυναίκες στην Ολλανδία. Και ε, ελπίζω όταν κάνουμε τον απολογισμό πεπραγμένων της Προεδρίας να μπορέσουμε να πούμε ότι σημειώθηκε πρόοδος. Μας περιμένει όμως σκληρή δουλειά. Πολύ πολλές μάλλον, Μπιόρκ ε, Ινφέλτ ε, αναφερθήκατε τα τραγικά περιστατικά της κολονίας και σε άλλες επίσης πόλεις της ε, Ευρώπης. Οι πολιτικές για τη χειραφέτηση και την ισότητα των ευκαιριών δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ποτέ ότι ολοκληρώνονται. Πάντοτε προκύπτουν νέες προκλήσεις, ε, θέτουμε νέους στόχους. Το Συμβούλιο ανησυχεί πάρα πολύ για την κατάσταση στην Κολονία και σε άλλες πόλεις ε, ήταν κατάφορη παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ε, των ίσων δικαιωμάτων των γυναικών αυτά που συνέβησαν και με αυτά τα περιστατικά θα αναδειχθεί σε προτεραιότητα αυτό το ζήτημα. Θα πρέπει να νιώθουν ελεύθερες, να μην φοβούνται οι γυναίκες ε, την κακοποίηση, να συμμετέχουν πλήρως στα κοινά με όλους τους πιθανούς τρόπους ε, και μέσω της νομοθεσίας ε, θα πρέπει να αγωνιστούμε γι' αυτό. Η βία, κυρία Λεγκρίπ, όποιες και αν είναι οι συνθήκες, όποια και αν είναι η φύση, όποιος και αν είναι ο υπέτειος, είναι επιλήψιμη πάντοτε και θα πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτά τα φαινόμενα. Το κράτος δικαίου δεν κάνει καμία διέκριση σε σχέση με την προέλευση, την κουλτούρα, τη θρησκεία, τις πεπιθήσεις των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε αυτή την διακριτική μεταχείριση για τους ανθρώπους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους. Θα πρέπει λοιπόν να αποφύγουμε αυτό το στίγμα κατά αυτή την ε, διακριτική μεταχείριση που υφίστανται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και να βρούμε αυτά που μας ενώνουν ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινέ λύσεις. Κατά τη διάρκεια της CSW στη Νέα Υόρκη το Μάρτι στα Ηνωμένα Έθνη θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε κάποια βήματα και νομίζω ότι θα είναι ε, ένα ζήτημα που θα συζητηθεί από τους ε, υπουργούς. Στη CSW σκοπεύουμε να θέσουμε αυτό το ζήτημα και φυσικά ασχολούμαστε επισταμένα με την εξέβρεση μιας λύσης. Έχουμε τη δήλωση του τρίου της Προεδρίας ε, το Δεκέμβρη που χάραξε το δρόμο και φυσικά ε, θα μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Κυρία Ίντφελτ, είναι επίσης σημαντικό να προστατεύουμε την ελευθερία των προσφύγων, τα ίσα δικαιώματα των γυναικών προσφύγων. Δεν θα πρέπει να διαχωρίζουμε αυτά τα ζητήματα προστασία των γυναικών από τη μία και από την άλλη πολιτική για τους πρόσφυγες. Ε, οι γυναίκες και τα κορίτσια ορισμένες φορές βρίσκονται σε λεπτότερη θέση και σίγουρα θα χρειαστούμε μια ε, λύση κατεπήγοντα μέτρα λόγω της ε, μεγάλης κρίσης που ζούμε αυτή τη στιγμή. Για τους ΛΟΑ δεν μπορώ να σας πω επειδή είμαι και υπουργό αρμόδια για τα ζητήματα χειραφέτηση ε, στην Ολλανδία, έχω αναπτύξει προγράμματα για την καταπολέμηση των φαινομένων βία κατά των γυναικών και των ΛΟΑΔΕ στα κέντρα υποδοχή προσφύγων. Αποδίδουμε τη δέουσα σημασία στο ζήτημα, λοιπόν. Κυρία Αρενά, ρωτήσατε γενικότερα για τη βία κατά των γυναικών. Έχει εκφράσει το Συμβούλιο τη δέσμευσή του για την πρόληψη και αποφυγή όλων των μορφών ουσιαστικά της βίας ε, κατά των γυναικών ε, και ε, υπέρ της εφαρμογής της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Το 2014 ήδη, αλλά και κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας, ε, κάναμε μια διάσκεψη σχετική και με το έγγραφο της Προεδρίας αναφερόμαστε στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και υποστήριξη των θυμάτων. Το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ συζήτησε και την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το, την περίοδο 2016 έως 2019 και όπως σας έλεγα η Σύμβαση Κωνσταντινούπολη έχει ιδιαίτερο ειδικό βάρος διότι αναγνωρίζονται γνωρίζονται αρμοδιότητες και εξετάζεται νομικός αντίκτυπος προσχώρησης. Εξετάζονται οι επιμέρους διατάξεις ε, και θα ρίνονται τα κράτη-μέλη να σημειώσουν πρόοδο ως προς ε, την εφαρμογή της σύμβασης. Αυτός είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να ε, αποδώσουμε την ιδιαίτερη σημασία σε αυτό το κέριο θέμα της βίας, κακοποίησης των γυναικών. Μιλήσατε για την ε, αυτοδιάθεση των γυναικών στο σώμα τους για τα δικαιώματα έκτρωσης. Φυσικά εξετάσουμε αυτά τα ζητήματα σε σχέση και με την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά έχουμε και την, το ψήφισμα του ΕΕ, όπως σας είπα, για τις γυναίκες και για την ειρήνη και το θέμα των φύλων ε, και η προστασία του σώματος των γυναικών έχουν ιδιαίτερη σημασία για την ενσωμάτωση της διάστασης ισότητας των δύο φύλων, κυρίως σε σχέση με την ομάδα υψηλού επίπεδου, φαίνεται πως σημασία δίνουμε σε αυτό το ζήτημα. Κυρία Ινφέλτε, για το σχέδιο δράσης για τους ΛΟΑΔ. Ξέρετε ότι η Επιτροπή το Δεκέμβρη παρουσίασε το σχέδιο δράσης ε, στο Συμβούλιο. Είναι ανεπίτρεπτη η διακριτική μεταχείριση κατά τον ΛΟΑΔ σαν παραβίαση των συνθήκων ε, και έχουμε ένα κατάλογο δράσεων για να εξασφαλιστεί η ισότητα των ε, ΛΟΑΔΕ για την ισότητα των δικαιωμάτων των δύο φύλων και των δικαιωμάτων των λοαδέ. έχει προετοιμαστεί ε, μία δήλωση η οποία αναμένεται να εγκριθεί το Μάρτι. Για το σεξουαλικό προσανατολισμό Φυσικά θα συνεχίσουμε την δουλειά που έχει γίνει ήδη για την οδηγία της ισότιμης μεταχείρισης. Απασχολεί εδώ και καιρό το Συμβούλιο το ζήτημα αυτό. Κυρία Ινφέλτ, επειδή είστε κι εσείς από την Ολλανδία, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά πως ε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας και σε όποιο επίπεδο μπορούμε για να καταπολεμήσουμε την ε, διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών ε, και τους ε, ΛΟΑΔ, κυρίως ενεργοποιώντας τον αρμόδιο οργανισμό στην Ολλανδία. για τα διοικητικά συμβούλια, για ε, τη θέση των γυναικών και εκπροσώπησή τους σε αυτά. Έχουν γίνει πάρα πολλά ε, σε σχέση με αυτή την οδηγία και στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και εκπροσωπώ εδώ την Προεδρία του Συμβουλίου. Παρ' όλα αυτά θέλω να τονίσω πως στην Ολλανδία η αναβάθμιση της θέσης των γυναικών σε μη εκτελεστικές θέσεις των διοικητικών συμβουλίων των επιχειρήσεων να συνιστά ύψιστη προτεραιότητα για μας και για να το επιτύχουμε αυτό έχουμε υιοθετήσει ένα θελοντικό στόχο για την εταιρική διακυβέρνηση. 5.000 περίπου επιχειρήσεις έχουν θέσει στόχο από πέρυσι λοιπόν τουλάχιστον σε ποσοστό 30% ε, αντρών και γυναικών στις ε, εκτελεστικές και μη εκτελεστικές θέσεις των διοικητικών συμβουλίων και αν δεν το επιτύχουν πρέπει να αιτιολογήσουν τη θέση τους σε μια αιτήσια έκθεση, ε, να αιτιολογήσουν γιατί δεν ε, εκπληρώθηκε ο προσδιορισμένος αυτός στόχος. Σας είπα ότι είμαι αρμόδια για τη χειραφέτηση στην Ολλανδία και πώς επιτυγχάνω τους στόχους μου. Ε, διορίζω πρέσβυρες στα, στα συμβούλια των επιχειρήσεων με στόχο την τόνωση, την αξιοποίηση των διεξιοτήτων των γυναικών σε ανώτερες θέσεις ε, του, ε, των διοικητικών συμβουλίων ε, και φυσικά συνεργαζόμαστε, κάτι που είναι καινούριο, και με τον ΟΑΕΔ στην Ολλανδία, με τον πρόεδρο του Οργανισμού Απασχόλησης. Να θυμίσω ότι το Δεκέμβρη στο Συμβούλιο υπήρξε μία μια αναστέλουσα μειοψηφία στο Συμβούλιο ε, και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας παρόλα αυτά για αυτή την οδηγία για την προσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Πάντως, ε, πρέπει να λάβουμε υπόψη τα όσα έχουν γίνει με αυτή την οδηγία. Χρειάζεται και προβληματισμός για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Οπότε, θα αφήσουμε αυτή την οδηγία στην επόμενη Προεδρία, εκτός και αν υπάρξει αλλαγή της θέσης του Συμβουλίου. Γι' αυτό το λόγο δεν θεωρήσαμε ότι συνιστά προτεραιότητα αυτή η οδηγία. Παρότι όμως κάποιος μπορεί να μην θεωρεί ότι συνιστά προτεραιότητα, μπορεί να εξακολουθεί να πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα για να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια, αλλά και για να μπορέσουμε να επιτύχουμε αυτή την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων. Ένα άλλο πιο γενικό ερώτημα κυρία Μπιόρκ για την περίοδο 2016 έως 2019 και τους στρατηγικούς στόχους. Αναφέρθηκα ήδη σε αυτό και φυσικά συνιστά θεμελιώδη αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στρατηγική ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το 2010 έως 2015 θα εκπνεύσει και η 22 κράτη-μέλη ζήτησαν την εκπόνηση νέας στρατηγικής. Στο τελευταίο έψκο συμβούλιο του Δεκεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης και κατά τη διάρκεια των συζητήσεων ε, πάρα πολλά κράτη-μέλη ε, τοποθετήθηκαν υπέρ αυτού του στρατηγικού σχεδίου για την επόμενη περίοδο. Εξέφρασαν όμως ε, την απογοήτευσή τους διότι δεν κατατέθηκε συγκεκριμένο σχέδιο δράσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι υποβαθμίστηκε σε επίπεδο απλής πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, χωρίς συγκεκριμένα μέτρα. Το Συμβούλιο κάλεσε στη συνέχεια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υιοθετήσει μια ανακοίνωση και μετά από αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προτίθεται το Συμβούλιο να εκδώσει και σχέδιο συμπερασμάτων. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει διαφωνία σε σχέση με αυτό, λοιπόν. Επόμενο ερώτημα, καλύτερη διακόπτη προεδρεύουσα. Ναι, δεν θα χρειαστώ πολύ χρόνο, λέει ο Υπουργός. Κυρία Γιούτο, δεν ξέρω παραφύρω το όνομά σας, έτσι το προφέρετε. Ε, αυτό είναι ένα θέμα της ε, Σλοβακικής ε, Προεδρίας και στην δήλωση με τη Μάλτα και τη Σλοβακία. Ήδη κάνουμε μια μνήμα, ναι, θα καταρτιστεί η έκθεση. Ίσως ξέρετε πως έχουμε αναλάβει τη δέσμευση για υπέρ της οικονομικής ανεξαρτησίας κατά πολέμηση στόχες ε, και της βίας κατά των γυναικών. Και αυτά τα ζητήματα είναι αλληλένδετα. Θα συνεργαστούμε στενά στα πλαίσια του τρίου της Προεδρίας για αυτά τα ζητήματα. Σας διαβεβαιώ πως το θέμα της καταπολέμησης φτώχειας θα μας απασχολήσει στους επόμενους μήνες. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να απήντηθε τουλάχιστον στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, ερωτήσεις. Ευχαριστούμε και ε, δεν μπορούσαμε να δώσουμε και άλλο χρόνο για του υπόλοιπου συναδέλφου να θέσουν ερωτήσει. Θα έχουμε άλλε ευκαιρίε να συζητήσουμε και έχουμε άλλο ένα σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να προσκαλέσω την κυρία Λάγκμπακ, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων, EIGE, e, για να συζητήσουμε τα μελλοντικά σχέδια και τι προγραμματιζόμενε δραστηριότητε του Ινστιτούτου.

Um, so we'll continue. Να συνεχίσουμε. Στην ημερήσια διάταξη έχουμε και άλλη παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων. Καλώ ορίζουμε την κυρία Λάγκμπακ, την διευθύντρια, και θα τη δώσω το λόγο για να μα παρουσιάσει τα βασικά αποτελέσματα και τι προγραμματιζόμενε δραστηριότητε, μάλλον τι δραστηριότητε που είχαν στο Ινστιτούτο το 2015. Ευχαριστώ πολύ, ε, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, Κυρίε και κύριοι. Σήμερα απευθύνομαι στο Κοινοβούλιο και στη δική σας επιτροπή και σε όλες τις υπόλοιπες σε αυτό το πλαίσιο με τις ε, απίστευτες καταστάσεις που ζει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συνεχιζόμενη κρίση, την μετανάστευση και τη διόγκωσή της ε, και την εσωτερική έλλειψη ασφάλειας. Όλα αυτά κλειδονίζουν τις κοινωνίες μας και είναι σημαντικό να μην τα δούμε ελαφρά την καρδία ε, ως θέματα που μπορούμε να τα λύσουμε με μια απλή σειρά προτεραιοτήτων. Όπως έδειξε ο δείκτης για την ισότητα των φύλων ε, στο Ινστιτούτο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει φτάσει μόνο στα μισά του δρόμου στην επίτευξη της ισότητας και τα στοιχεία τα μετρούμε μόνο από το 2005. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις δομές για την λήψη αποφάσεων ε, στο χώρο εργασίας το ίδιο και τα πράγματα επιδεινώνονται και όλα αυτά ε, δυστυχώς ε, επιτείνονται από τις μορφές βίας, ψυχολογικής, σωματικής και σεξουαλικής όπως ακούστηκε σήμερα και στις διάφορες ερωτήσεις που τέθηκαν. Επίσης τα στερεότυπα, οι προκαταλήψεις ενισχύονται συχνά και από άλλα προβλήματα οι πρόσφυγες που φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές. Όλοι ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και αυτό προσθέτει στην άκρα δεστησία αυτού του τμήματος του πληθυσμού. Στη δουλειά του το Ινστιτούτο προσπαθεί να φωτίσει από κάποια από τα προβλήματα αυτά, να τα εξετάσει από την πλευρά της κατάρτισης πολιτικής και να βοηθήσει τους πολιτικούς ευθύνοντες με τις ειδικές μας γνώσεις, ώστε οι πολιτικές που θεσπίζονται να μπορούν να ωφελήσουν και τις γυναίκες και τους άντρες. Αλλά ταυτόχρονα να προστατεύσουν και τους πλέον ευάλωτους. Να επικεντρωθώ λοιπόν σε μερικούς τομείς, τέσσερις, οι οποίοι αντικατοπτρίζουν το τι κάναμε το 2015 που θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το 2016. Πρώτα απ' όλα το θέμα της φτώχειας αναφέρθηκε από αρκετές ερωτήσεις από τις βουλευτές της ερωτήσεις τους. Η Ευρώπη σήμερα έχει 65 εκατομμύρια γυναικών και 58 εκατομμύρια ανδρών που ζουν ε, με τον κίνδυνο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Όταν μιλάμε για τη γυναική διάσταση στη φτώχεια, το φύλλο είναι συχνά ένα παράγον που ε, ενισχύει τα στατιστικά αυτά δεδομένα, ιδίως σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες για παράδειγμα, κάθε ένα δευτερόλεπτο ένα μόνο γονέα με δύο παιδιά αντιμετωπίζει τον κίνδυνο τη φτώχεια. Σήμερα στην Ευρώπη και 88% αυτών των ε, μόνων γονέων είναι γυναίκε παιδιά που μεγαλώνουν σε φτωχέ οικογένειε, ε, που κινδυνεύουν από την φτώχεια, αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα όταν μεγαλώσουν ω ενήλικοι και δεν καταφέρουν να σπάσουν τον κύκλο τη φτώχεια. Αυτό λέει, ε, λένε οι έρευνε. Όταν η φτώχεια είναι κάτι που το γίνει βίωμα, συνήθω αποτελεί μια μόνιμη παρέα για τη ζωή ε, του ανθρώπου. Είναι λοιπόν ένα θέμα που αφορά τι γυναίκε και σε μικρέ και σε μεγάλε ηλικίε, όμω οι ηλικιωμένε αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο ε, λόγω των εντυνόμενων ανισοτήτων στο τέρμα προ το τέλο του κύκλου ζωή. Το ίδιο και το μισθολογικό χάσμα, οι πισπαλεί συνθήκε εργασία, οι διακοπέ λόγω των ε, φροντίδων που συχνά αναγκάζονται να παρέχουν οι γυναίκε οδηγούν και σε συνταξιδοτικά κενά και μεγαλύτερο κίνδυνο η απειλή από τη φτώχεια όταν μια γυναίκα φτάνει σε μεγάλη ηλικία. Οι μετανάστες είναι επίσης ένας ευαίσθητο, ένα ευαίσθητο μερίδιο του πληθυσμού γιατί και αυτοί ζουν στα όρια τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού. Χρειάζονται περαιτέρω μελέτε για να αποκαλύψουμε το πρόβλημα σε όλη του την έκταση, καθώ και τη φύση τη όλη κατάσταση, ιδίω υπό το φω των σημερινών μεταναστευτικών ροών και τη αυξανόμενη πίεση προ τα κάτι μελη όλο ιδιαίτερο, για να σχεδιάσουν βιώσιμα μέτρα για την κοινωνική ένταξη όσων μείνουν και ενσωματωθούν στι ευρωπαϊκέ κοινωνίε. Κατόπιν αιτήματο τη επικείμενη Σλοβακική προεδρία το ΕΙΓΕ ετοιμάζει μία έκθεση για την φτώχεια, όπω αναφέρθηκε σήμερα και από την Υπουργό, για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα αναλύσουμε πώς η φτώχεια αλληλοσχετίζεται με την ηλικία, με την εθνικότητα, την ε, προέλευση, την εθνοτική και την ε, οικογενειακή κατάσταση. Επίσης πώς επηρεάζει η κρίση. Η έκθεση που θα απευθύνεται στη Σλοβακική Προεδρία θα συμπληρώνεται από μια συλλογή καλών πρακτικών για μέτρα παρακολούθησης που μπορεί να αποκαθιστούν τη διάσταση αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ως το τέλος του 2016 επίσης η έκθεση αυτή θα στηρίξει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου και τα μέτρα που πρέπει να αναλυθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα συνεχιστεί δράση στους τομείς όπου οι ανισότητες και η φτώχεια συναντώνται σε συνδυασμό με τον παράγοντα της ισότητας των φύλων και των ε, διασταυρούμενων ανισοτήτων. Ε, επίσης, λόγω της επικείμενης προεδρίας, και αφού μας το ζήτησε η Μαλτέζικη Προεδρία, ε, είδαμε την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και από τη σκοπιά της απασχόλησης και σχεδιάζουμε να εκπονήσουμε έκθεση που θα αναλύει πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε τις δεξιότητες των γυναικών για να καλύψουμε ανάγκες στον εργασιακό χώρο. Οι μακρόχρονες απουσίες, η έλλειψη ευκαιριών, η πρόσβαση στην εκπαίδευση λόγω κοινωνικο-οικονομικών δυσκολιών, όλα αυτά μπορεί να οδηγήσουν τις γυναίκες και να τις παγιδεύουν σε χαμηλόμιστες θέσεις ή να παραμένουν διαρκώς σε επαγγελματική φτώχεια. Ένας δεύτερος τομέας και σε αντίθεση με τη φτώχεια ή βία κατά των γυναικών δεν εξαρτάται ούτε από την εθνικότητα, την ηλικία, ούτε από την προέλευση του καθενό, αν είναι μετανάστευση ή όχι. Ε, αφορά τα κοινωνικά στρώματα και όλε τι εκφάνσει του βίου. Η βία κατά των γυναικων δεν εξαρταται δυστυχώ έχει εμποτίσει κοινωνικέ συμπεριφορέ, προκαταλήψει και πρότυπα που ακούγονται και αναφέρονται σήμερα στι κοινωνίε μα και δεν μπορούν δραστικά να αντιμετωπιστούν χωρί να, διαγραφούν τα, τα στερεότυπα περί φύλων. Οι νοοτροπίες αλλά και η στάση της, στην βία κατά των γυναικών δεν έχει να κάνει μόνο με την αναζήτηση ενόχων αλλά και με την ε, περιορισμένη παρέμβαση χρειάζεται, υποστήριξη των θυμάτων. Χρειάζεται οι αρχέ να είναι ευαισθητοποιημένε, να επιτρέπει την δικτύωση των θυμάτων μεταξύ του. Ένα παράδειγμα, έγινε μία έρευνα στην Πολωνία, 80% των ερωτηθέντων ε, συμφώνησαν ότι δεν υπάρχει βιασμός ε, μεταξύ συζύγων ή συντροφών. Οι νέοι στην Κύπρο έλεγαν ότι 15% των αγοριών θεωρούσα ότι μπορεί ένα αγόρι να απαιτήσει από το κορίτσι του να δίνεται έτσι ή αλλιώς. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι να δει κανεί με κάποια απόσταση τα πρότυπα αυτά που ισχύουν σε εμά και τι αξίε μα, ιδίω όταν αφορά το φαινόμενο τη μετανάστευση. Το ίδιο με το πώ θα φωτίσουμε τι διάφορε εκφάνσει τη βία ε, κατά των γυναικών και των στερεοτύπων που τις πλήττουν. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια εύρωστη βάση δεδομένων. Οπότε το Ινστιτούτο θα συνεχίσει να βελτιώνει τα δεδομένα που συλλέγει για τη βία κατά των γυναικών, συγκεντρωνόμενο στην συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων και υποστηρίζοντα τα κάθε μέλη στην εκπλήρωση των, των υποχρεώσεών του για την παρακολούθηση και την εφαρμογή τη οδηγία για τα δικαιώματα των θυμάτων και ταυτόχρονα για την κύρωση τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Για το πλαίσιο των μετρήσεων ο τομέας των δικτών συγκριτικής αξιολόγησης, ιδίως για τη βία, θα χρησιμοποιεί όλους τους ε, αξιόπιστους δείκτες που συστηματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταμετρούν ε, τις διατάσει του φαινόμενου αυτού και τις επιπτώσεις από τη δράση μας για τη βία κατά των γυναικών. Ο γυναικείος γενετικός ακροτεριασμός ε, βασίστηκε στην αντιμετώπιση του σε έναν οδηγό βαθμιαίο που εντοπίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από την κλήτορη δεκτομή και το Ινστιτούτο μας παρέχει συνδρομή στα κάτι μέλη για την υλοποίηση της θετικής αυτής. Η βία κατά των γυναικών είναι ένα ζωτικό θέμα που πρέπει να δούμε στο πλαίσιο και της σημερινής μεταναστευτικής κρίσης. Είναι πολύ άριθμες ε, οι εκθέσεις που καταγράφουν τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών στην γυριά Ευρώπη πρέπει οι υποδομές μας για την ε, υποδοχή ή εγκαταστάσεις για και τα προγράμματα ένταξης να λάβουν την απαραίτητη στήριξη και να υπάρχει πρόσβαση όλων στην οικονομική περίθαλψη. Αυτό λοιπόν που θα επιδιώξουμε να γίνει είναι να γίνει μια καλή ανάλυση των ε, προβλημάτων που προκύπτουν για τους πρόσφυγες και τους οτούντες άσυλο σε σχέση με την οικονομική περίθαλψη. Έπειτα η επαρκής ανταπόκριση στις νέες, στα νέα προβλήματα απαιτεί προσαρμογή και των ε, διαδικασιών λήψη αποφάσεων. Πρόσφατα η έκθεση μας για τη Λουξεμβουργιανή Προεδρία έδειξε ότι ενώ κάποια πρόοδο επιτελέστηκε σε πολλού τομεί, ιδίω στην πολιτική, Υπάρχουν αποδεκτικά στοιχεία που δείχνουν ε, σαφώς ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις δομές λήψης αποφάσεων, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές. Οι άντρες ακόμη υπερέχουν στις κεντρικές τράπεζες, τα Υπουργεία Οικονομικών και τα Διοικητικά Συμβούλια σε όλη την Ευρώπη. Ένας στους 25 γενικούς διευθυντές είναι γυναίκα. Στις 28 κεντρικές τράπεζες μόνο ένας από τους πρόεδρους είναι γυναίκα στην Κύπρο και μόνο δύο γυναίκες είναι υπουργοί οικονομικών στη Ρουμανία και τη Σουηδία. Καθώς ο κόσμος ετοιμάζεται για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Ρίο και τους παραολυμπιακούς εκεί, η σχετική κουβέντα γίνεται πολύ επίκαιρη η εκπροσώπηση των γυναικών στα σώματα λήψης αποφάσεων και στους αθλητικούς συλλόγους της Ευρώπης είναι πραγματικά περιθωριακή. Για να τονίσουμε αυτό το πρόβλημα και με την αφορμή της Παγκόσμιας ημέρας των γυναικών θα οργανώσουμε ένα διεθνές σεμινάριο για την ισότητα των φίλων στα ε, αθλήματα, στα σπορ στο Βίλνιους. Και έπειτα οι αποτελεσματικές πολιτικές για την ισότητα των φύλων δεν μπορεί να υπάρξουν απομονωμένες. Η ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων, το gender mainstreaming, ήταν σημαντική διάσταση του έργου μας. Φέτος είχαμε μια πλατφόρμα πλήρως αναπτυγμένη για το θέμα αυτό, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όλους τους χρήστες, πολιτικούς υφήνοντες, με εργαλεία, κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές για την ευθυγράμμιση τη διάσταση τη ισότητα των φύλων σε όλου του τομείς πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, από την ενέργεια και τι υποδομέ μέχρι τι κοινωνικέ υποθέσει, την απασχόληση και τον πολιτισμό. Επίση, αναπτύσσουμε ένα εργαλείο ανάλυση για να συλλέγουμε εμπειρικά δεδομένα για την ευαισθησία σε σχέση με την ισότητα των φύλων και το γιατί συμβαίνει στα κοινοβούλια. Τα κοινοβούλια με τα πρακτικά τους πλαίσια για την αυτο αξιολόγησή τους και το κατά πόσον επικρατεί μια ε, νοοτροπία στον εργασιακό αυτό χώρο για να δέχονται τα κοινοβούλια τις ανάγκες των γυναικών και ως φροντιστών. Η διάσταση αυτή στα κοινοβούλια, όπως η λειτουργία το ίδιο του κοινοβουλίου ως σώματος ή η σύνθεση, η θέση των γυναικών στο θεσμικό όργανο, οι συνθήκες εργασίας τους και οι πρακτικές που χρησιμοποιούν αλλά και οι πολιτικές, οι νόμοι που παράγουν τα κοινοβούλια και που μπορεί να ωφελούν την κοινωνία ευρέως, όλα αυτά θα πρέπει να ε, οδεύουν στο στόχο προστασίας της ερώτας των φίλων θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα συνεχίσουμε να είμαστε κεντρικός ε, συνομιλητής του Κοινοβουλίου στα θέματα ισότητας των φύλων. Ελπίζουμε να παραμένουμε αφοσιωμένος και χρήσιμος συνεργάτη σας καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα έχει συζήτηση για τα λόγια απόψεων. Αν έχετε ερωτήσεις και θέλετε να τις κάνετε, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ, με τη σειρά. Η κυρία Μίλη, η Βάνα μετά. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, πολύ ε, εκτενής και εξαντλητική η αναφορά σας και η έκθεση. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στενή συνεργασία με τον οργανισμό σας. Έχω να σας κάνω μία πρόταση. Ως εισηγήτρια για το gender mainstreaming θα προσκαλούσα ε, το ΕΕ και να έχει συνεργασία μόνιμη και πάγια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια δομή φιλόδοξη και προσβλέπουμε στη δική σας συνεργασία. Να σας δώσω και παραδείγματα που χρειαζόμαστε την υποστήριξη στην κατάρτιση υπαλλήλων και βοηθών η στενή συνεργασία με το δίκτυο για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές, το λεγόμενο gender mainstreaming και να μας βοηθήσετε να μειώσουμε την απόσταση και το χάσμα που χωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ξέρουμε ότι τρέχει ένα δικό σας πρόγραμμα, ένα έργο ε, για ευαισθητοποίηση ε, σε θέματα φύλου και θα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να μάθουμε από εσά, να αντιγράψουμε θέλετε το πρόγραμμά σας, να διδαχθούμε από τις εμπειρίες σας. Αυτό είναι το αίτημα που θα είχα να σας απευθύνω και θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας απόψεις σχετικά. Η κυρία Βάνα, ευχαριστώ πολύ. Εγώ μιλάω γερμανικά και θα σας παρακαλούσα να βάλετε τα ακουστικά σας γιατί θέλω να φερθώ σε ειδικού τομείς και δεν ξέρω τους όρους σε άλλες γλώσσες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη εντύπωση ε, μου έκαναν αυτά που άκουσα και το φάσμα των δραστηριοτήτων που καλύπτεται είναι πάρα πολύ καλά τα όσα μας λέτε και για τη βάση της λήψης των αποφάσεών μας, όχι μόνο σε αυτή την Επιτροπή και σε άλλες Επιτροπές. Το είπε και η κυρία Μίλνα υπάρχουν ε, και άλλες εκθέσεις και το gender mainstreaming παίζει ρόλο σε όλες τις επιτροπές και σε όλες τις εκθέσεις. Θέλω να ρωτήσω κάτι εγώ ε, για την περιφερειακή πολιτική. Είμαι στην ε, Περιφερειακή Επιτροπή Αρμόδια για θέματα φύλου και εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την πολιτική των επενδύσεων και πώς κατανέμονται τα κονδύλια από τα διευθυντικά ταμεία ή από το νέο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στην περιφέρεια. Έχω λοιπόν την εξή ερώτηση. Είναι πάρα πολύ λίγα τα στοιχεία που έχουμε για την ε, πολιτική ισότητα στην περιφέρεια, στην Ήπεθρο και τις επιπτώσεις. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς έχετε τέτοια στοιχεία και αν ναι, έχουν να κάνουν με την περιφέρεια, έχουν να κάνουν με τις αστικές περιοχές, με την Ήπεθρο, γιατί και η ε, Ολλανδική Προεδρία εστιάζει σε αυτό. Και μια άλλη ερώτηση. Συμφωνώ πολύτως Αυτά που είπατε για τη βία κατά των γυναικών, αυτό δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με την ε, καταγωγή ή την προέλευση. Βλέπουμε τον Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα που δείχνει ε, τι διαστάσεις έχει η ενδοοικογενειακή βία σε όλη την Ευρώπη ή στο κοινωνικό περίγυρο της γυναίκας. Είναι τρομακτικά τα στοιχεία. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το βλέπετε. Δεν θέλω η συζήτηση να γίνει αυτή για ε, λόγους ή υπό ένα πρίσμα μεταναστευτικό ή προσφυγικό. Δεν είναι καθόλου κάτι τέτοιο. Και επίση έχετε ποσοτικά στοιχεία ε, και στοιχεία που να επιτρέπουν τις ποσοτικές ε, συγκρίσεις. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι που έχει να κάνει με την ποιοτική διάσταση. Έχετε συγκρίνει το ποινικό δίκαιο ε, των διαφόρων κρατών μελών και πώς τιμωρεί ε, κάποια εγκλήματα βία σεξουαλικά κατά των γυναικών. Εγώ είμαι από την Αυστρία και τώρα έχουμε πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση του ποινικού δικαίου και γίνεται μεγάλη συζήτηση για την σεξουαλική παρενόχληση, την παρενόχληση σε δημόσιο χώρο, το βιασμό και άλλα σεξουαλικά εγκλήματα. Το δικό μας ποινικό δίκαιο θεωρείται πολύ καλό και παρόλα αυτά δεν θα κάλυπτε ε, ε, ικανοποιητικά ε, περιπτώσεις τέτοιων κακουργημάτων όπως αυτά που είδαμε πρόσφατα στην Κολονία. Και ακριβώς επειδή εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και τις διάφορες οδηγίες, έχετε κάνει καμιά ποιοτική σύγκριση του ποινικού δικαίου από χώρα σε χώρα και πώς τιμωρεί τέτοιου είδους εγκλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Με μεγάλη μας χαρά ετοιμάζουμε μια διεξοδική βάση δεδομένων για τα θέματα αυτά μια πλατφόρμα για την ευθυγράμμιση της διάστασης της ισότητας των φύλων. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται το Κοινοβούλιο και προκειμένου να περατώσουμε την αποστολή δεδομένων προς το Κοινοβούλιο. Διότι βεβαίως και θέλουμε να ε, έχουμε ρεαλιστική αντιμετώπιση εν ώψη των διαβουλεύσεων. Αυτό είναι και για μας χρήσιμο. Για τα δεδομένα. Δεν άκουσα. Παρακολουθούσα τη διερμηνία. Δεν κατάλαβα εάν θέλετε δεδομένα για συγκεκριμένες περιφέρειες, γενικώ για την ισότητα των φύλων, για όλων των ειδών του τομείς που, που αφορά η ισότητα των φύλων. Ε, τώρα ολοκληρώνουμε και πολύ σύντομα θα ξεκινήσουμε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων στατιστικών. Θα καταγράφουμε ό,τι διατίθεται για να μπορούν εύκολα να τα χρησιμοποιούν οι χρήστες. Θα γίνεται ένα login ε, σε ένα μόνο σημείο και θα συγκεντρώνει κανείς αμέσως όλα τα χρήσιμα στοιχεία για την ισότητα των φύλων. Ανακατηγορία, βλέποντας τι διατίθεται και από το Eurostat και από κάποιους από τους φορείς μας, φορείς μας, τους οργανισμούς μας. Θα μπορεί κανείς λοιπόν να τα βρει εύκολα ή θα μπορεί να γίνει και μια έρευνα εκ μέρου σα εφόσον στείλετε συγκεκριμένο αίτημα. Πάντως, αυτή η βάση δεδομένων θα επικαιροποιείται συστηματικά. Μόλις έχουμε νέα δεδομένα θα τα συμπεριλαμβάνουμε και θα προσπαθούμε συστηματικά να ε, ενημερώνουμε για την προσθήκη δεδομένων. Ξέρουμε ότι αυτό υπάρχει στη Eurostat, είναι κάτι που ήδη προβλέπεται και τώρα συζητάμε και με την Επιτροπή των Περιφερειών, με το Συμβούλιο της Ευρώπης, Προσπαθούμε να έχουμε μια ενιαία βάση λοιπόν για όλες τις περιπτώσεις και να τα συμπεριλάβουμε. Για τη βία κατά των γυναικών. Ε, είναι κάτι που το ξεκινήσαμε πέρσι και νομίζω τον ε, Δεκέμβριο είχαμε μια εκδήλωση στο Κοινοβούλιο για το πώς τιμωρείται η βία και πώς ε, διαμορφώνεται η κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Έχουμε μια έρευνα με διοικητικές ε, πηγές για τη βία κατά των γυναικών και δύο εκθέσεις. Μία για, την, ε, για το νομικό σύστημα, το νομοθετικό σύστημα κάθε κάποιους μέλους και τι προβλέπει για τη βία κατά των γυναικών. Τα αναλύουμε και έχουμε καταρτήσει και πίνακες για να δούμε τι συμβαίνει σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή, ποια είναι ποιες είναι οι διάφορες ποινές, τι μέτρα ισχύουν Εάν θέλετε να σας στείλουμε το link για να τα δείτε. Επίσης, συζητήσαμε με αφορμή την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης το θέμα αυτό στο επίπεδο της αρμόδιας επιτροπής θα πρέπει να δούμε πώς τα κράτη-μέλη υλοποιούν τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και αυτό και μέσα από τη δική μας δουλειά. Είχαμε μια πρώτη συζήτηση για αυτήν τη συνεργασία και για την ποιοτική διάσταση που ε, την αναπτύσσει εκτενώς η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Είναι κάτι που και αυτό που να το αναλύσουμε. Επίσης, περατώνουμε τώρα το πλαίσιο μετρητών για την ισότητα των φίλων στην περίπτωση της βίας και προσπαθήσαμε για πρώτη φορά να δημιουργήσουμε ένα συμπληρωμένο δίκτυ με την ποιοτική διάσταση για τη διάκρατα των γυναικών ε, που μπορεί να συσχετιζόταν με την ισότητα των φύλων ώστε να δούμε πώς υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις βίας, περιπτώσεις βίας που καταγράφονται και πώς αυτές παρουσιάζονται εκ των υστέρων. Μας ενδιαφέρει εδώ όλος ιδιαίτερος η ποιοτική διάσταση, ε, η σεξιστική συμπεριφορά, Όλες οι μορφές εξάσκησης βίας θα αναλυθούν, αλλά αυτά θα έχουν διατεθεί μέχρι το τέλος της χρονιάς φέτος. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις, δεν ξέρω, άλλος κανείς θέλει να ρωτήσει τίποτα, όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για όλες τις προφορίες που μας δώσατε. Έχουμε τίποτα στα διάφορα, έχει κανείς κανένα διάφορο, όχι. Ωραία, καλώς ραντεβού στις 17 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ, χαίρετε.